So, good afternoon, ladies. Καλό σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Για, για να αρχίσουμε. Καταρχάς, η πρόεδρος, η κυρία Ματσόνη, θα καθυστερήσει επειδή έχει μία συνάντηση με Ιταλό Υπουργό και γι' αυτό θα προεδρεύσω εγώ προσωρινά που να έρθει η πρόεδρος μας. Το πρώτο θέμα είναι η υιοθέτηση του η έγκριση του Ιδίου ημερησίας διατάξεως. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε λίγα λεπτά πριν από την ψηφοφορία αύριο. για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε καλά το έργο μας και να έχουμε ένα περιθώριο συζήτησης, να τα πούμε μεταξύ μας. Αύριο. Η πρόεδρος. Ναι, ωραία. Ας μην απαντήσω γιατί η κυρία Ματσόνη θα χειριστεί τις εργασίες μας ε, αύριο και το χρόνο πριν από την ψηφοφορία. Εκείνη είναι υπεύθυνη. Λοιπόν, σημείο 1. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί με δύο βασικά ντοσιέ, σε οποία είναι πρώτον η παρουσίαση της μελέτης για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη από τον Κρίστιαν Νόιμπαουρ και τον Χούμπερτ Ράισιγκερ. Θα γίνει μια παρουσίαση με διαφάνειες της μελέτης αυτής και ο κύριος Ιτούργαης είναι εισηγητής του θέματος αυτού και θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο θέμα σήμερα είναι συζήτηση του προϋπολογισμού και περικοπές του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Ε, αυτό το θέμα και οι συνέπεια των περικοπών στη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων προσθέθηκε ως κατεπήγον θέμα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπαλτσάνη για τον προϋπολογισμό του 2012 και θα είναι παρούσα. Εκπρόσωποι των ετούντων θα είναι παρόντες επίσης όπως και στελέχη από τα διοικητικά συμβούλια των ε, σχολείων και εκπρόσωποι των ενώσεων γονέων και μαθητών. και διευθυντές των Ευρωπαϊκών Σχολείων. main Οι συντονιστές εν συνεχεία θα συνεδριάσουν στις 5.30 μετά από τις συζητήσεις των δύο προαναφερθέντων βασικών θεμάτων που έχουμε σήμερα. 5.30 με 6.30 λοιπόν συντονιστές. Αύριο η κυρία Ιώτοβα θα λείπει και θα γίνει συνεχεία στο σημείο 12 μια προκαταρτική προφορική έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στη Βουλγαρία. Τώρα, αναφερόμενοι για αύριο είναι εξή. Σημείο 13, ο κύριος Ρούσεφ, εξ ονόματος της εταιρείας Bull Limited, σχετικά με την κατάχρηση πόρων 15 Ήμπορα Μπερνάλ 16 κυρία Καμίλα Κλίν Πέτερσεν 17 Μπιέλαβα για τα αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί όσον αφορά τώρα τον ε, αναφέροντα για την διακίνηση στην Ιρλανδία, έχει αποσυρθεί. Ε, 19, Peter Brown, 20, Deboni, ε, ε, αντιμονοπολιακοί κανόνες. Η 18 λοιπόν έχει αποσυρθεί. Στο Β, τα πρακτικά λοιπόν της προηγούμενης συνεδρίασης έχουν ε, διανεμηθεί. Ε, έγκριση των πρακτικων 20-24 Μαΐου, σημείο 3 ανακοινώσει του Προέδρου και αυτό έχει διανεμηθεί. Δεν ε, έχουμε λάβει παρατηρήσεις και σχόλια, οπότε θεωρούνται και κρυμμένα. Σημείο 4 είναι τα διάφορα. Η γραμματεία δεν έχει λάβει προτάσεις από το σημείο διάφορα. Πάει και αυτό, το διευθετήσαμε. Και ξέχασα στην αρχή να σας αναφέρω ότι η μερίσια διάταξη έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις γλώσσες, στα συστηρίδες και στα ντοσιέ των μελών. Αυτά ως προς τις ε, ανακοινώσεις του Προέδρου, της Προέδρου μάλλον. Και ας αρχίσουμε τώρα τις εργασίες μας. Ο αναφέρον για την ε, αναφορά ως προς το περιβάλλον δεν είναι παρόν και θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Σαμπρό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε. Συναντηθήκαμε λοιπόν για να συζητήσουμε την ε, αναφορά της κυρίας Κατιούσε Ευερλιγκέρη Ιταλικής Ιθαγένειας σχετικά με την διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στις επαρχίες του Σαλέρνο, του Αβελίνο και του Μπενεβέντο στην Ιταλία. Πρόκειται για την υπαριθμό 387 κάθετο 2008. Η αναφέρουσα καταρχάς μας είχε ε, δώσει πολύ λεπτομερή τεκμηρίωση όσον αφορά ε, την υποστήριξη των λεγόμενων της. Γνωρίζετε βεβαίως ότι το Ταμείο Φεντέρ μπορεί να συγχρηματοδοτήσει πολιτιστικού περιβάλλοντος δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και της διατήρησης της ιστορικής κληρονομιάς και της φυσικής ε, κληρονομιάς. Από την πλευρά του, ο ΦΕΟΓΑ τμήμα εγγύησεων και προσανατολισμών μπορεί να συγχρηματοδοτήσει παρόμοιες παρεμβάσεις για την ε, ανακαίνιση χωριών και για την προστασία της κληρονομιάς της υπαίθρου. Όμως, βάσει της αρχής της ε, ε, μοιρασμένης διαχείρισης, οι αρχές διαχείρισης στα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνες για την επιλογή και την υλοποίηση αυτών των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Όσον αφορά το ΦΕΝΤΕΡ, τον Ιούνιο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με την επαρχία της ε, Καμπανίας και συγκεκριμένα ε, με τους τοπικούς υπεύθυνους του εκεί επιχειρησιακού σχεδιασμού ε, των προγραμμάτων που αφορούσαν στη χρηματοδότηση του ΦΕΝΤΕΡ 2006-2007 έτσι ώστε να διακριβώσουν κατά πόσον ε, υπήρξε συγχρηματοδότηση βάσει των καταγγελιών της αναφέρουσας. και αν η υλοποίηση του προγράμματος προχωρούσε κανονικά. Νομίζω ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν ήδη λάβει μία πρώτη απάντηση από την πλευρά μας και εν πάση περιπτώσει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πρόσφατες εξελίξεις και ότι θα είμαστε σε θέση ε, πολύ γρήγορα να σας αποστείλουμε περαιτέρω ενημέρωση για αυτές τις νέες εξελίξεις. Οι τοπικές αρχές όντως μας απήντησαν όσον αφορά το ΦΕΝΤΕΡ την 23η Μαΐου του 2011 και μας πληροφόρησαν ότι δύο ε, ε, σχέδια είχαν συγχρηματοδοτηθεί με τις ε, τοπικές αρχές του Κασάλμπο και του Κασταλβέκιο. Το πρώτο βάση του ε, προγραμματισμού 2000-2006 ε, και επίσης το δεύτερο όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα ε, του 2007-2013 ε, και με πρόκειται χρηματοδότηση ύψους 1,7 δις. Εκατομμυρίων, συγγνώμη. Ε, τα προγράμματα αυτά αφορούν την ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ε, επαρχία του ε, Αβελίνο ε, και στην Διαχειριστική Επιτροπή είναι παρόντα και μέλη της τοπικής αρχαιολογικής εφορίας. Επομένως, η αναφέρουσα για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί στις εθνικές της αρχές. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση του ΦΕΟΓΚΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 26η Μαΐου του 2011 ήρθε σε επαφή με τις ε, αρχές διαχείρισης που είναι υπεύθυνε για την υλοποίηση μέτρων ε, ανάπτυξης της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένου και του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της υπαίθρου, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι και στην προκείμενη περίπτωση οι ευρωπαϊκοί πόροι χρησιμοποιήθηκαν σωστά και σύμφωνα με τις ε, ε, μορφές παρέμβασης που η αναφέρουσα ε, περιλαμβάνει στην αναφορά της. Είχαμε απάντηση την 31η Μαΐου, σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια μέτρων συγκεκριμένων ε, του επιχειρησιακου προγράμματο προγράμματος 2000-2006. Και επίσης, την 5η Ιουλίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, οι περιφερειακές αρχές μας πληροφόρησαν ότι κατά την άποψή τους οι εργασίες έλαβαν χώρα με τρόπο φυσιολογικό ε, και με στόχο μάλιστα την βελτίωση αγροτικών περιοχών ε, και την διατήρηση είτε ε, χωριών είτε γενικότερα του τοπίου της υπαίθρου. Επίσης, το Ιταλικό Υπουργείο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Πολιτισμού έδωσε την άδειά του για εργασίες στην τοποθεσία την οποία ε, καταγράφει η αναφέρουσα. Επομένως, οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει γνώση για οποιαδήποτε ανομαλία ε, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου γενικότερα. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να υπογραμμίσει ότι κατά την άποψή της η εκτέλεση των εργασιών αυτών δεν αφορούν δική της αρμοδιότητα, δεν εμπίπτουν ε, σε πεδίο αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις που έλαβε και ότι ενδεχομένως ε, η αναφέρουσα ε, θα έπρεπε να ε, στραφεί προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ε, να, να ρωτήσω τον Πιέτρο Μόρα δεν ξέρω αν βρίσκεται εδώ πέρα η κυρία Νικουλή επίση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιε ερωτήσει αυτή τη στιγμή, κάποιε παρατηρήσει. Θα ήθελα πάντω να του δώσω τον λόγο, εφόσον το επιθυμούν. Καλημέρα σα. Πιέρ Νικόλα Πρέμολη λέγομαι και μπορώ να μιλήσω Ιταλικά, βεβαίω μπορείτε. Εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής, ε, ε Περιφερειακής Πολιτικής, ε, κυρία Αντιπρόεδρε σε σχέση με αυτά που μόλις ακούσαμε από την συνάδελφό μου. Μπορώ να σας πω, να προσθέσω μάλλον κάποια ιδιαίτερα στοιχεία. Είναι κρίμα που η δόκτωρ Κατιούσε Βελιντζέρη δεν είναι εδώ, γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε έτσι μια συνολικότερη αντιμετώπιση της αναφοράς που από ό,τι καταλαβαίνω αφορά ε, την καταστροφή κάποιων ε, ιδιαίτερης αξίας ε, στοιχείων και που αποτελεί προφανώς πλήγμα για την πολιτιστική κληρονομιά. Κοιτάξτε, βάσει των παρελθόντων και υφισταμένων κανονισμών ε, για το, που διέπουν μάλλον το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα τα οποία αφορούσαν την περιοχή της ε, καμπάνιας 2000-2006 και 2007-2013, και που μερικά προγράμματα που πέφτουν στο μετέχμιο των δύο περιόδων. Παρόλα αυτά, λέγω, δεν μας δίνεται καμία δυνατότητα παρέμβασης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εμείς μπορούμε να παρέμβουμε μονάχα σε περίπτωση που δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Επομένως, όταν οι τοπικές αρχές εγκρίνουν, και όχι οι Κομισιόν, εγκρίνουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για μια αρχαιολογική ε, ή πολιτιστική τοποθεσία, οι ίδιες ε, οι αρχές, οι διαχειριστικές, θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσον οι αρχές ε, οι οποίες ακολουθούνται είναι αυτές ε, οι οποίες ε, είχαν εξαγγελθεί τον, στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Δηλαδή, εάν ο διαγωνισμός έλεγε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν 10 θέσεις εργασίας μόνιμες και έχουν δημιουργηθεί 10 εποχικές, τότε τα πράγματα δεν είναι σωστά. Όμως, θα μπορού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως κάνει κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους οικονομικούς ελέγχους ε, για να δει εάν όντως υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη και δεν έχουν γίνει σεβαστά κάποια κριτήρια. Στα κριτήρια πάντως δεν περιλαμβάνεται ε, καθόλου στην προκείμενη περίπτωση η κατεδάφιση ή η καταστροφή κάποιων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ε, αυτό ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να επαγρυπνά έτσι ώστε ε, να μην καταστρέφεται η πολιτιστική κληρονομιά ή να χρησιμοποιούνται ε, οι σωστές τεχνικές συντήρησης. Στην προκείμενη περίπτωση λοιπόν που αν δεν κάνω λάθος πρόκειται για καταστροφή τμήματων του κάστρου Πινιατέλη δεν μπορούμε εμείς σαν Κομισιόν να παρέμβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πρέμολη, μάλλον ο κύριος Πρέμολη, παρακαλώ κύριε Πρέμολη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, εγώ λέγομαι Πιέρο Μόρα, από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και ε, παρεμβαίνω σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από τον ΦΕΟΓΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2000-2006. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που η συναδελφό μα σας αποσαφήνισε. Να προσθέσω όμως ενδεχομένως ότι βεβαίως μα ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, και προσέχουμε ε, πάρα πολύ και παρακολουθούμε οποιασδήποτε περιπτώσεις ε, φτάνουν στην προσοχή μας και στι οποίε υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία για κακή διαχείριση ή κακή χρήση των πόρων του Ταμείου και ε, βεβαίως ε, μπορούμε να παρέμβουμε και διατηρούμε την δυνατότητα παρέμβασης με ενδεχόμενη απέτηση επιστροφής των καταβληθέντων πόρων σε περίπτωση ανομαλίας. Αυτό θέλω να σας το διασφαλίσω και επίσης να σας πω ότι λαμβάνοντας υπόψη ε, όλες τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν και εδώ και όλες τις πληροφορίες τις οποίες ε, είχαμε εμείς, ε, βάσει λοιπόν όλων αυτών επιβεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο χρηματοδοτήθηκε βάσει του μέτρου ανακαίνησης χωριών και στοιχείων τοποθεσιών της υπαίθρου φαίνεται λέω να μην υπάρχει καμία ανομαλία ή κακή χρήση των χρημάτων. Πάντως διατηρούμε την προσοχή μας συγκεντρωμένη στην περίπτωση αυτή αν χρειαστεί και αν προκύψουν κάποιες εξελίξεις. Θέλει κάποιος άλλος, λέει η Πρόεδρος, να πάρει το λόγο. Η κυρία Ούκεν, παρακαλώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Όντω εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Ουσιαστικά δεν απαγορεύει κανείς σε χώρε να καταστρέφουν την πολιτιστική του κληρονομιά. Είναι μέρος της δημοκρατίας και αυτό. Ωστόσο θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε κάνει μια αξιολόγηση περιβαλλοντικής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει και με την πολιτιστική κληρονομιά. Περιλαμβάνεται στα πλαίσια της οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε μια τέτοια αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει λάβει χώρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εμπλέκονται και οι πολίτες σε αυτή την αξιολόγηση. Και άλλωστε αυτό προβλέπεται, όπως σας είπα, και από την ίδια την οδηγία. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, σας λέω όχι. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάνει κάποια μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Όντως θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι τέτοιο, υπό συγκεκριμένων όμως προποθέσεων. Η κυρία θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι προβλέπεται στην οδηγία και η μελέτη αυτή η επιπτώση που θα μπορούν να έχουν κάποια έργα, κάποιες εργασίες στην πολιτιστική κληρονομιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε δίκιο. Γίνονται όμως και κάποιες μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όντως σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε επιδείνωση της πολιτιστικής ε, κληρονομιάς. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις για το ζήτημα αυτό. Αν όχι, μπορούμε να περάσουμε στην ε, δεύτερη αναφορά. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Επομένως, κλείνουμε αυτή την αναφορά. Έτσι δεν είναι, λέει ο Πρόεδρος. Εφόσον δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, άλλες παρατηρήσεις, άλλα σχόλια ή ερωτήσεις, μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά και να περάσουμε στην επόμενη Ευρωπαϊκά Σχολεία. Η κυρία Όκεν, ναι, αλλά κλείνοντας την αναφορά αυτή θέτουμε και ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. can reopen <laughs> this point. Πρόεδρος. Κυρία Όκεν, μάλλον. Θέλω απλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει στα όσα υπόθηκαν στη συνεδρίασή μας. Μα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ήδη, λέει η Πρόεδρος. Δεν σας αρκούσε προφανώς η απάντηση αυτή, κυρία Όκεν. Όκεν. Μα δεν αρκεί να λέμε απλώς ότι δεν έγινε κάτι. Πρέπει να λάβει χώρα η μελέτη αυτή σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόεδρος, νομίζω όμως ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο τουλάχιστον. Αυτό που το οποίο προβλέπεται από την Επιτροπή μας είναι ότι θα δούμε τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτή την αναφορά. Περνάμε όμως στην επόμενη αναφορά ευρωπαϊκά σχολεία. Με συγχωρείτε λέει η Πρόεδρος. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος, δεν είχα το σωστό έγγραφο μπροστά μου. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κρίστιαν Νόιμποϊερ να κάνει μια παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας σήμερα. Το όνομά μου είναι Christian Neubauer και ο συνάδελφός μου Hubert Reisinger. Προερχόμαστε από την περιβαλλοντική υπηρεσία της Αυστρίας και συντάξαμε τη μελέτη αυτή βάσει συγκεκριμένων αναφορών που είχαν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην εξέταση των κυρίων των βασικών προβλημάτων και στη διατύπωση ε, συστάσεων και προτάσεων για το μέλλον. Τα επόμενα, τα επόμενα 20 λεπτά λοιπόν θα σας παρουσιάσω αυτή την μελέτη για τα βασικά σημεία. Καταρχάς, ε, θα σας κάνω μια ανασκόπηση των αναφορών που εξετάσαμε. Πήραμε 101 αναφορές και ε, σημειώσαμε τις ε, τρεις βασικές προβληματικές πτυχές. Όπως σας είπα λοιπόν, 101 αναφορές μελετήθηκαν ενδελεχώς για, τη, για την έρευνα που κάναμε και κάλυψαν το διάστημα 2004-2010. Την πρώτη αξιολόγηση που κάναμε, προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε τις αναφορές σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια και Εν συνεχεία κάναμε μία νομική αξιολόγηση για να επισημάνουμε τις, πιο, τις διατάξεις που ήταν οι πιο σχετικές, τις πιο σχετικές διατάξεις μέσα στις οποίες εμπίπτουν αυτές οι αναφορές. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα, τους πίνακες αυτούς, ορισμένα από τα επιλεγή γέντα, ορισμένα τα επιλέξιμα κριτήρια και την ομαδοποίηση που κάναμε των αναφορών αυτών ε, βάσει του, του, της γενεσιουργού αιτίας της αναφοράς. Τα περισσότερες αναφορές λοιπόν είχαν ως στόχο την ε, παροχή αδείας και τις, ε, την, διάφορες διαδικασίες σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 50, μία. 48 είχαν ως στόχο την ε, λειτουργία μιας υπάρχουσας εγκατάστασης και 25 την λειτουργία διαχείρισης αποβλήτων. Εν συνεχεία, ομαδοποιήσαμε τον, ε, τη μορφή των εγκαταστάσεων, τον τύπο των εγκαταστάσεων όπως ξέρετε, οι περισσότερες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι χωματέρες. Δεκαεφτά ήταν αποτεφρωτές, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. 13 ήταν ε, άλλης μορφής ε, διαχείριση αποβλήτων και μόνο τέσσερις αναφορές αναφέρονταν σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής. Ένα άλλο κριτήριο ήταν η νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν οι αναφορές. Ε, βασικά ήταν έξι ευρωπαϊκές οδηγίες ε, στις οποίες αναφέρονταν οι περιπτώσεις αυτές. Ήταν οι πιο δηλαδή επίκαιρες ε, οδηγίες αυτών των αναφορών. 44 αναφορές αναφέρονταν στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, 43 στην οδηγία για τις χωματορές, Εν συνεχεία άλλες οδηγίες όπως η μελέτη επιπτώσεων ε, και άλλες συναφείς οδηγίες. Εκεί είχαμε 32 περιπτώσεις αναφορών. 15 βασίστηκαν στην οδηγία της IPPC και 5 ε, στην οδηγία αποτέφρωσης αποβλήτων. Εν συνεχεία, βλέπετε το είδος. Τι έγινε. But I think the next chart will be better. So it's only this chart. You can also... Ε, βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά ο τελευταίος πίνακας, αλλά υπάρχει, έχουμε τυπώσει και την ε, ε, παρουσίαση αυτή για να δείτε καθαρά τα στοιχεία και τους αριθμούς. Ένα άλλο λοιπόν κριτήριο ήταν η μορφή, ο τύπος των αποβλήτων, επικίνδυνα, επικίνδυνες ουσίες, επικίνδυνα απόβλητα, στερεά απόβλητα, τοξικά απόβλητα, μη επικίνδυνα απόβλητα, κοινοτικά, στερεά απόβλητα κλπ. Εκτός λοιπόν από την ομαδοποίηση των αναφορών βάση κριτηρίων, κάναμε και μία αξιολόγηση νομικής φύσεως προσπαθήσαμε να εξετάσουμε λεπτομερώς τις έξι αυτές οδηγίες που ανέφερα και να τονίσουμε ποιες διατάξεις, ποια μεμονωμένα άρθρα είναι τα σχετικά, τα συναφή, αυτά δηλαδή τα οποία έχουν άμεση σχέση με την αναφορά. Η πιο ε, δημοφιλής οδηγία, ας το πούμε έτσι, ήταν η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα του 2006 κάθετος 12 Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 4. Από αυτές τις 101 αναφορές, 25 αναφορές ε, βασίστηκαν στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006, κάθετος 12. Ε, πρέπει να σας πω ότι αυτή η οδηγία πλαίσια είναι παλιά. Και αναθεωρήθηκε το 2008. Αναφέρω, όταν λέω λοιπόν οδηγία πλαίσιο για τα, για τα πόβλητα, ε, αναφέρομαι στην παλιά, το 2006. Έτσι λοιπόν, το άρθρο 4 αναφέρθηκε σε 25 αναφορές. διότι αναφέρεται ακριβώς σε, στη χρησιμοποίηση μεθόδων που δεν βλάπτουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Όπως βλέπετε και το άρθρο 9 αναφέρθηκε και το άρθρο 10, 13 φορές Και αυτά τα άρθρα 9 και 10 αναφέρονται στην εγκυρότητα των αδειών λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε επισημένοντας ποιες αναφορές αναφερόντουσαν σε συγκεκριμένα άρθρα των συγκεκριμένων έξι οδηγιών. και βλέπετε ακριβώς σε ποιες οδηγίες και σε ποια άρθρα επικεντρώνονται οι αναφορές. Εν συνεχεία, κάναμε μια γεωγραφική ε, ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων ανάλογα με τη μορφή τους, στο βορρά της Ευρώπης, αν βλέπετε, χοντρικά δηλαδή υπάρχουν λιγότερες χωματερές, ενώ στο νότο και νότιο δυτικά υπάρχουν αρκετές, αρκετοί αποτεφρωτές ε, και βλέπετε ακριβώς που υπάρχουν τα προβλήματα ε, στις χωματερές, ε, στους αποτε... στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ε, στις βιομηχανικές διαδικασίες διάθεσης αποβλήτων κλπ. Δεν είναι μόνο δηλαδή η παλιά ευρωπαϊκή κοινότητα ή οι καινούργιες χώρες, αλλά υπάρχει μια διασπορά προβλημάτων. Εκτός λοιπόν αυτή την γεωγραφική αξιολόγηση, διαπιστώσαμε που ότι πάνω από το 90% των αναφορών ε, αναφέρονταν σε τοπικές συνθήκες και ένα ελάχιστο ποσοστό σε ένα εθνικό επίπεδο και μόνο μία σε υπερεθνικό επίπεδο. Τρεις, λοιπόν, προβληματικές τρεις προβληματικοί τομείς διαπιστώθηκαν. Ο πρώτος προβληματικός τομέας είναι η μη συμμόρφωση σε ε, διαδικασίες που επιτρέπονται. Ο, ο δεύτερος τομέας προβληματικός είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω ακατάλληλης λειτουργίας και ο τρίτος τομέας προβλημάτων είναι ελλείψεις και ε, ακατάλληλες, ε, ακατάλληλος σε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το λόγο έχει ο κύριος Ρέιζιγκερ. Θα ήθελα να σας δώσω και εγώ κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη γραφική αυτή παράσταση. Βλέπετε εδώ πέρα από ποιες περιοχές προέρχονται οι περισσότερες αναφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και με την παρουσία, με την παρουσία χωματερών. Επίσης βλέπουμε στη γραφική αυτή παράσταση και άλλες μεθόδους, όπως για παράδειγμα καύση αποβλήτων. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πολλές χωματερές, ακολουθούν στη συνέχεια κάποιες εγκαταστάσεις, κάποιες μονάδες αποτέφρωσης. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε εδώ πέρα είναι ότι ε, δεν έχουμε αναφορές από κάποιες βόρειες χώρες, από το Βέλγιο μέχρι τη Φιλανδία. Τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο δεν έχουν υποβληθεί αναφορές όσον αφορά την ε, διαχείριση των αποβλήτων. Τι εξήγηση μπορεί να δοθεί στο φαινόμενο αυτό. Μια εξήγηση είναι ότι οι χώρες αυτές είναι τόσο προηγμένες στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν διάφορα συστήματα διαχείρισης, ανακύκλωσης και συλλογής ε, των αποβλήτων, συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεχομένως οι χώρες αυτές να έχουν ήδη και κάποια συστήματα πρόληψης, ελαχιστοποίησης, παραγωγής ε, αποβλήτων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις και επομένω υπάρχουν και λιγότερες διαφορές όσον αφορά την υποδομή με τις άλλες γειτονικές τους χώρες. Πρόκειται για τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη παράδοση όσον αφορά την εμπλοκή του δημοσίου τομέα. Επομένω, οι χώρες αυτές ε, έχουν τις απαραίτητες υποδομές ε, και κατά αυτόν τον τρόπο εξηγείται ενδεχομένω η θετική αυτή εικόνα που έχουμε στι βόρειε χώρε. Η αρνητική πλευρά μας των πραγμάτων είναι ότι στι χώρε αυτέ η δαπάνη διαχείριση των αποβλήτων θεωρείται υψηλότερη από ότι στις χώρες εκείνες οι οποίες εξαρτώνται από χωματερές. Ας περάσουμε έτσι στην επόμενη διαφάνεια, στην πρώτη δηλαδή περίπτωση, στην οποία αναφερόμαστε στις αναφορές εκείνες, τις οποίες θεωρούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες μη συμμόρφωσης. Η πρώτη αναφορά έχει να κάνει με την χωματερή Σουχοντόλα, την βασική χωματορή της Σόφιας στην Βουλγαρία. Η χωματερή αυτή έκλεισε σε μια πρώτη φάση και στη συνέχεια χωρίς να έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου άνοιξε πάλι. Ήταν η μόνη επιλογή ουσιαστικά που υπήρχε για τη διαχείριση αποβλήτων στην περιοχή. Στη συνέχεια έχουμε την χωματερή Πεζινόκα, στην Πρατισλάβα της Σλοβακίας. Εκκρεμεί εδώ πέρα μία προσφυγή στο δικαστήριο, όπου το ανώτατο δικαστήριο και το συνταγματικό δικαστήριο δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν για το αν ε, η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου είναι πιο σημαντική ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του διαχειριστή της χωματερής αυτής που έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη συνέχεια έχουμε τις χωματερές του Γραμματικού και της Κερατέας χωματερές και ιδίω στην Ελλάδα και έχουν επιλεγεί προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα διαχείρισης ε, αποβλήτων της περιοχής των Αθηνών, ενώ η τέταρτη αναφορά έχει να κάνει με τη χωματερή Pathhead Query του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ε, και εκεί φάνηκε ότι ε, είχαν εντοπιστεί προβλήματα στην μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Τα κριτήρια επιλογής τα οποία ακολουθήσαμε είχαν ως στόχο να επιλέξουν τις πιο ουσιώδεις αναφορές. Επιλέξαμε λοιπόν τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα ανάμεσα στην ε, βασική αστική περιοχή της χώρας και τις γειτονικές περιοχές. Εστιάσαμε λοιπόν δηλαδή στις ε, πιο προβληματικές περιοχές για τις οποίες έχουν υποβληθεί αναφορές. Αυτό το οποίο εντοπίσαμε στις αναφορές αυτές είναι ότι η απουσία υποδομών οδηγεί είτε σε παράνομη διάθεση αποβλήτων ή στην ανάγκη δημιουργίας μιας εναλλακτικής λύσης. Η σύστασή μας λοιπόν είναι να κινηθεί κανείς ανωδικά στην αναγκη δημιουργιας μιας συναλλακτικής λυσης η συσταση μας λοιπον αυτή της διαχείρισης των αποβλήτων όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση όπου θα πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των απορριμμάτων, αλλά και οι απαραίτητες υποδομές για την ανακύκλωση, διαχείριση των απορριμμάτων αυτών. Θα μπορούσε να γίνει αυτό με την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά την ανακύκλωση των απορριμμάτων και θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με την ε, χορηγία επιπλέον πόρων και κονδυλίων. Παράλληλα θα μπορούσαν να επιβληθούν και υψηλότερε κυρώσει για την παράνομη διάθεση των απορριμμάτων. Σε ορισμένε επίση περιοχέ ε, θα μπορούσε να βελτιωθεί το όλο σύστημα καταγραφής των παράνομων απορριμμάτων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι ε, οι αρμόδιοι φορείς είτε δεν ε, ενεπλάκησαν είτε επενέβησαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις περιοχές αυτές. Αναφέρομαι στις περιοχές εκείνες όπου ε, απαιτούνται νέες υποδομές, ακόμα και αν πολλές φορές δικαστήρια στις χώρες αυτές έχουν αποφασίσει ότι πολλές φορές οι χωματορές αυτές δεν συνάδουν με την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία και πάλι υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι στην απόφαση αυτή και πολλές φορές βλέπουμε ότι ο τοπικός πληθυσμός δεν επιθυμεί την κατασκευή νέων υποδομών. Η σύστασή μας λοιπόν στην περίπτωση αυτή είναι να ακολουθήσουμε το θετικό παράδειγμα των βόρειων χωρών προκειμένου τα εμπλεκόμενα μέρη να επεμβαίνουν πολύ γρηγορότερα, να δημιουργούν την απαραίτητη ικανότητα και υποδομή, προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο θα διεξάγει τόσο τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, που θα είναι σε θέση να ακολουθήσει επίσης τα βέλτιστα παραδείγματα που έχουμε από άλλες χώρες, Επίσης, ε, σε ορισμένε ε, χώρες ο φορέας ε, παροχής, ο οικονομικός φορέας που διαχειρίζεται τις χωματερές αυτές είχε υποστηρίξει ότι ακολουθούνται τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια προκειμένου οι χωματερές αυτές να γίνουν αποδεκτές. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει τα αυστηρότερα δυνατά κριτήρια και να επιβάλλει επίση και μια ελάχιστη γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στι χωματερέ και τι περιοχές όπου κατοικούν οι πολίτε. Επίση, θα πρέπει να υπάρχουν ε, διάφορα συστήματα διασφάλιση του περιβάλλοντο, συστήματα για παράδειγμα που θα μπορούσαν να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο και που θα μπορούσαν να προβλέπουν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνιστούμε επίσης να υπάρχει μια μεταφορά γνώσεων προς τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτές οι χώρες δηλαδή θα πρέπει να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν τα καλύτερα δυνατά διδάγματα που έχουν οι χώρες που ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές. Όσον αφορά τώρα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που απορρέουν ε, από τις ε, δραστηριότητες ε, των, των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τέσσερις συγκεκριμένε, ιδιαίτερα δύο αναφορές. Εδώ τα κύρια προβλήματα είναι ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, εκπομπές οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες. Θα ήθελα τώρα να περάσω στην ε, επικέντρωση στα προβλήματα και τις ε, συστάσεις μας. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο απομονώσαμε είναι ότι πολλές φορές η αδειοδότηση δεν είναι σωστή και δεν έχει γίνει βάση των ε, διεθνών νόμων. Ας πούμε στο άρθρο 4 της οδηγίας σχετικά με την συμμόρφωση των αδειοδοτήσεων προς την οδηγία φαίνεται ότι δημιουργεί πρόβλημα. Η σύσταση που δίνουμε εδώ είναι ότι θα πρέπει να δοθούν και στις εθνικές αλλά κυρίως στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να δοθούν, λέω, διοικητικές δυνατότητες, γιατί αυτές οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ως νομοθετική επιλογή μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να, υπάρξουν, να υπάρξει επιπλέον εξειδίκευση ε, των ε, αδειών που θα αφορά και το περιεχόμενο και τη διάρκεια και την ε, συχνότητα κτλ. Και βεβαίως να πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν και ε, οι επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να γίνονται επιτόπου επιθεωρήσεις. Άλλες επιλογές θα ήταν ενδεχομένως ε, κάτι που έχουμε ήδη προαναφέρει, ε, να υπάρξει δηλαδή να δοθούν μεγαλύτερες δυνατότητες παρέμβασης στις τοπικές αρχές, το είπαμε και στις ε, προτάσεις που κάνουμε για τις νομοθετικές επιλογές και επίσης ε, να δοθεί και κάποια ε, καθοδήγηση. Το επόμενο πρόβλημα το οποίο έχουμε απομονώσει είναι ότι οι άμεσες εκπομπές από τις διαδικασίες αυτές δεν ελέγχονται πάντα και δεν εποπτεύονται με τρόπο ικανοποιητικό. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν διαρκείς μετρήσεις. Ε, θα πρέπει να ενδυναμωθεί το σύστημα μετρήσεων, κυρίως δε ε, μετρήσεις των κεντρικών εκπομπών, καθώς επίσης και όλων των παραμέτρων σε όλη τη διάρκεια των διεργασιών. για όλα αυτά τα συστήματα ε, διαχείρισης ε, αποβλήτων η ε, προσπάθεια ελέγχου των εκπομπών είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό τι μπορούμε να πούμε σαν νομοθετικές επιπτώσεις είναι ε, σε εθνικό επίπεδο να καταγραφούν οι ελάχιστες ε, απαιτήσει όσον αφορά τις μετρήσεις εκπομπών και όσον αφορά τις ε, παραμέτρους όλων των διεργασιών των διαφόρων μορφών διαχείρισης αποβλήτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά και σε όλες τις ε, περιπτώσεις ε, θα πρέπει ε, να καθοριστούν σαφείς και λεπτομερείς προϋποθέσεις. Το επόμενο πρόβλημα που διαπιστώσαμε είναι ότι μερικές φορές ε, όταν ε, στις ε, διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων δεν φτάνουν τα σωστά απόβλητα, τότε δημιουργούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια κριτήρια, δηλαδή θα πρέπει να αποσαφινιστούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων έτσι ώστε κάποια ανεπιθύμητα στοιχεία ή ανεπιθύμητες ουσίες να παραμείνουν έξω από το σύστημα διαχείρισης ε, ε, αποβλήτων. Επίσης θα πρέπει να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν ε, συστήματα ελέγχου, δοκιμών και δειγματοληπτικών ελέγχων. Πολύ σύντομα τώρα, να συνεχίσω. Σε αυτή την περίπτωση της, ε, του τρίτου προβλήματος εξετάσαμε διάφορες αναφορές από την περιοχή της Καμπάνια και στο Γήθιο, στη Νότια Πελοπόννησο στην Ελλάδα, λιγότερες περιπτώσεις, όπου το πρόβλημα είναι περιφερειακό και αυτό συμφωνεί και με τις διαπιστώσεις που είχαμε κάνει προηγουμένως, ίδιες συστάσεις ε, και ίδιες επιλογές, όπως και με τις περιπτώσεις 1 και 2. Δεν θέλω να τα επαναλάβω λοιπόν. Η περίπτωση 3, καμπάνια και γήσιο, έχει τις ίδιες προτάσεις και συστάσεις όπως οι δύο προηγούμενες. Απλώς συνοπτικά να πω ότι Υπάρχουν δυνατότητα θα βελτιωθεί το σύστημα σε ορισμένες χώρες και να βρεθούν ε, ή να δημιουργηθούν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων που δεν θα οδηγήσουν σε παράπονα και αναφορές. Ε, αυτές ε, οι περιπτώσεις, ας πούμε οι καλές περιπτώσεις ε, γίνονται όταν ζητεί, γίνεται προηγούμενη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Ε, στην συνεχεία να μην υπάρχουν τριβές. Η σε ευχαριστώ πολύ. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία ήταν αυτή. Και τώρα έφτασε η ώρα για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια. Θα δώσω... Όπως καταρχάς το λόγο στην Κομισιόν και στην Επιτροπή, στη Λίμπε, στην ε, Α, είμαι και εγώ σκιώδη εισηγήτρια από τους, ΛΥΜΠΕ, από τους φιλελεύθερου, για ένα συναφέ θέμα. Λοιπόν, όπως είπε και η, προ... η τελούσα χρέη Προέδρου, δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ε, είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τμήμα διαχείρισης αποβλήτων. Δεν είχαμε καιρό μέχρι τώρα να εξετάσουμε τη μελέτη αυτή. Το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι να σας παρουσιάσω ορισμένα προκαταρτικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι καλή, είναι θετική. Η, η αξία της έγκυται στο ότι ξεπερνάει την οπτική γωνία των αναφορών και ε, βασίζεται σε, μια ευρύτερη, σε ένα ευρύτερο πεδίο μελέτης και αναφέρεται σε συστάσεις που θα οδηγήσουν στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και υπό αυτό το πνεύμα είναι πολύ καλή μελέτη. Ε, τέσσερα πέντε σημεία βασικά θέλω να θίξω διαβάζοντας σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση Βλέπω ότι γίνονται ορισμένε προτάσεις νομικής ε, φύσεως, αλλά πιστεύω γενικά ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρύτατο πλέον. Και ε, πιστεύω ότι αυτό το νομοθετικό ε, πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων είναι ευρύτατο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ε, ε, η γεωγραφία, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων και των προβλημάτων όπου αναφέρονται οι αναφορές, πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις περιπτώσεις 6 και 7 που αναφέρονται στην έκθεση. αναφέρθηκε από τους ομιλητές ένα μοντέλο διανομής, διασποράς μάλλον, των προβλημάτων βορρά-νότου. Αυτή η σύγκριση των προβλημάτων δείχνει ότι σε κάτι μέλη που έχουν μία υψηλής ε, τεχνολογικής ε, ποιότητα συστήματα βελτίωσης ε, διαχείρισης αποβλήτων υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές οι αναφορές αυξάνονται γεωμετρικά στα κράτη-μέλη όπου ο ρυθμός ανακύκλωσης, διαχείρισης, αποτέφρωσης κλπ. είναι πάρα πολύ χαμηλός και όπου βασικά χρησιμοποιούνται χωματερές. Αυτή η επιλογή της χωματερής πράγματι είναι μια επιλογή η οποία από τεχνικής απόψεως είναι ξεπερασμένη, σαφής, σαφώς και δημιουργεί ακριβώς τα περισσότερα προβλήματα στην ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτή την άποψη θα ήταν χρήσιμο να τονιστεί στη μελέτη η σημασία της νέας οδηγίας διαχείρισης αποβλήτων και ε, τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει για τη βελτίωση του συστήματος. είναι αυτή η οδηγία αναφέρεται συγκεκριμένα σε στόχους ανακύκλωσης μέσα στο πλαίσιο της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων και επίσης της ε, σαφείς ε, διατάξεις για το διαχωρισμό των απορριμμάτων και τον διαχωρισμό των αποβλήτων. Πιστεύω ότι με αυτές τις σαφείς διατάξεις θα σημειωθεί μια ε, χειροπιαστή βελτίωση στη διαχείριση των αποβλήτων γενικά. Η μελέτη τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης συγκεκριμένων, ε, του συγκεκριμένου δυναμικού στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εφόσον βεβαίως τοπικές αρχές ή περιφερειακές αρχές είναι οι αρμόδιες για τη διαχείριση των αποβλήτων. Όμως πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να είχε αναφέρει καταρχάς το ρόλο των, του, εθνικών δικαστών ιδίω σε θέματα τοπικής αντίδρασης όπου προτείνεται η εγκατάσταση μιας μονάδας διαχείρισης αποβλήτων και Επίσης, να αναφερθεί ε, στις εθνικές ε, δικαστικές ε, διαδικασίες που έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση αυτών των αντιδράσεων. Επίσης, είναι σαφές ότι εμείς στην Κομισιόν δεν πρέπει να αντιγράψουμε ένα εθνικό σύστημα επιθεωρήσεων, αλλά η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να, να γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις υπηρεσίες της Κομισιόν να παρακολουθούν τις ε, συστημικές αποτυχίες ε, του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ε, και ε, του νομικού πλαισίου. Στις σελίδε 44 44-45 αναφέρονται οι, δια, οι αποτεφρωτές και οι εγκαταστάσεις καύσης, αποτέφρωσης των αποβλήτων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφέρεται αυτό το δίκτυο και πιστεύουμε ότι η ανάλυση αυτή στην ε, μελέτη θα βοηθήσει να ξεπεραστούν ορισμένες παρανοήσεις και παρερμηνίες ε, του όλου θέματος ε, της αποτέφρωσης των αποβλήτων. Στην Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι ότι η καύση, η αποτέφρωση πρέπει να παίξει έναν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων και πρέπει να αναπτυχθεί αυτός ο τρόπος να διευρυνθεί. Αυτή η βούλησή μας είναι σαφέστατη. Δεύτερον, στην Κομισιόν είμαστε πεπισμένοι ότι ε, η επατέφραση των αποβλήτων είναι απόλυτα ασφαλής μέθοδος και δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις, ε, έχει, δεν έχει επιπτώσεις ε, στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Και τέλος, θα αναφερθώ ε, στην οτροπία αυτή του μη ρίχνετε τα σκουπίδια ε, στη δικιά μου αυλή. Ή μάλλον εγώ να, μη να ρίχνω τα σκουπίδια μου στις αυλές των άλλων. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στη διαχείριση και στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Ε, είναι σαφές ότι αυτό το απαιτεί και η κοινωτική νομοθεσία. Όμως, ε, ταυτόχρονα είναι σημαντικό ναι, να αναγνωρίσουμε ότι οι κάτοικοι και οι τοπικοί ε, φορείς έχουν και αυτοί να λέγουν. πρέπει να ακούγονται ε, και πολλές φορές ε, η τοπική αντίδραση από τους κατοίκους μπορεί να μπλοκάρει και να παρεμποδίσει την ε, λειτουργία, την, την κατασκευή μιας εγκατάστασης και να δημιουργήσει σημαντικότατα προσκόμματα στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε βεβαίως ε, και την ε, ε, υπηρεσία η οποία ανέλαβε και συνέταξε, εκπώνησε και παρουσίασε την μελέτη αυτή. Τουρκάνης πρώτα και μετά ο επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτήν την ε, ε, μελέτη η οποία μας φάνηκε πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Έγιναν και ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα σχόλια και η μελέτη αυτή εμπλουτίζει την έκθεση αυτή την οποία θα παρουσιάσω ως εισηγητής με τη βοήθεια βέβαια σκιωδών εισηγητών από άλλες πολιτικές ομάδες. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα προς τους συντάκτες της μελέτης γιατί θέλω να αποσαφηνίσω κάποια σημεία. Καταρχάς, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την δημόσια συμμετοχή, τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα όσον αφορά την διαδικασία αδειοδότησης για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης και πώς θα καταφέρουμε να πείσουμε το κοινό να αποδεχθεί περισσότερο τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Έχετε κάποια άποψη γι' αυτό. Δεύτερον, θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα στους ε, φορείς παροχής των υπηρεσιών αυτών, τους δημόσιους φορείς και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκούμενους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζει ποιε είναι οι δικέ σα απόψει για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Τρίτον, όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, οι κανόνε που ακολουθούμε ισχύουν από το 1985 και ισχύουν για πολλού δημόσιου και ιδιωτικού φορεί. Αυτό το βλέπουμε στο παράρτημα 1 και στο παράρτημα 2. Στο παράρτημα 1 βλέπετε όλα τα προγράμματα αυτά για τα οποία είναι υποχρεωτική η περιβαλλοντική μελέτη και στο παράρτημα 2 έχουμε ένα κατάλογο προγραμμάτων όπου η περιβαλλοντική μελέτη εναπόκειται σε απόφαση που θα πάρει το κράτος μέλος. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική. Ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά την ιδέα να γίνουν ακόμα πιο δεσμευτικέ και υποχρεωτικέ οι μελέτε αυτέ, δηλαδή η αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου να είναι υποχρεωτική για όλα τα σχέδια τα οποία προβλέπονται στα δύο αυτά παραρτήματα. Have... Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Όκεν, σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Είπατε ότι στην, στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης μάλλον δεν έχετε αρκετές αναφορές από τις βόρειες χώρες. Πολύ ωραία. Αν όμω θέλετε πραγματικά να ανταποκριθείτε σε αυτή την ιεράρχηση που έχετε κάνει, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, για παράδειγμα, στη δικιά μου τη χώρα, τη Δανία, αποτεφρώνουμε τα πάντα. Τα πάντα, εκτός βέβαια από τα βιολογικά απόβλητα. Και προβλέπεται αυτό σε όλη την αλυσίδα παροχής ενέργειας. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια ενδεχομένως να έχετε πολύ λίγες αναφορές η αποτέφρωση γίνεται με ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια μόλυνση από τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια της αποτέφρωσης αυτής, στα πλαίσια της καύσης, και με πολλών λογιών ε, υλικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές χώρες βέβαια, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ιεραρχία στην οποία αναφερθήκατε. Δεν ε, ασχολούνται ιδιαίτερα με τις μεθόδους ανακύκλωσης και πολλές φορές επειδή ε, έχουν να κερδίσουν οικονομικά από τη στάση τους αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν εσείς στη δική σας μελέτη το έχετε λάβει αυτό υπόψη σας. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υποβληθούν αναφορές προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε αν μια χώρα συμμορφώνεται ή όχι με τις ε, υποχρεώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην οδηγία. Και αν έτσι τα πράγματα, τότε αυτοί που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό θα πρέπει πραγματικά να υποβάλουν αναφορές για το ζήτημα αυτό. Γιατί Σαφώς ακόμα και στις βόρειες χώρες θα μπορούσαν να ακολουθηθούν διαφορετικές μέθοδοι. Έχουν παγιωθεί απλώς κάποιες μέθοδοι αυτή τη στιγμή. Στην ε, Κοπεχάγη, για παράδειγμα, μάθαμε ξαφνικά ότι ε, υπήρχε ένας τρόπος να καταφέρουμε να ξεφορτωθούμε κάποια προβληματικά μας απόβλητα. Έμαθα βέβαια στη συνέχεια ότι δεν το κάνουν αυτό προκειμένου να βοηθήσουν εμά του πολίτε, αλλά ενδιαφέρονταν για τα απόβλητα αυτά, γιατί ουσιαστικά θα παρήγαγαν ενέργεια με αυτά. Επομένω είχαν και αυτοί να κερδίσουν από την διαδικασία αυτή. Όσον αφορά λοιπόν την εμπλοκή των πολιτών, θα ήθελα να την τονίσετε περισσότερο στην μελέτη σας. Είχα πάει και στην καμπανία της Ιταλίας, ασχολούμαι και με το ζήτημα των χωματερών της Ουγγαρίας και το πρόβλημα το οποίο έχω εντοπίσει τελικά είναι ότι οι πολίτες δεν εμπλέκονται καθόλου στην όλη διαδικασία δημιουργίας ενός συστήματος βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων. Αν δεν ε, περιλάβετε στις μελέτες σας αυτές τους πολίτες, δεν θα καταφέρετε ποτέ να έχετε επιτυχία. Παρακαλώ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και τους ε, κυρίους που παρουσίασαν αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα μελέτη. Οι αναφορές ε, που σχετίζονται με τα απόβλητα και τη διαχείριση των ε, αποβλήτων βεβαίως βρίσκονται στο κέντρο των εργασιών της Επιτροπής μας διαπιστώνουμε ε, ότι βεβαίως υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι αυτοί είναι καλοί, αλλά κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά ε, την εφαρμογή τους. Διαφορετικά δεν θα είχαμε τόσες πολλές αναφορές. Ήδη έγινε κατανοητό μέσω της ε, εργασίας σας, έγινε κατανοητό το τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, βλέπουμε ότι οι νόμοι ευρωπαϊκοί υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πολλές ελλείψεις. Άρα πρέπει να βρούμε ε, τις ελλείψεις αυτές, ε, να τις ταυτοποιήσουμε. Διαπιστώσαμε επίσης ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα χρηματικό. Δεν είναι δηλαδή τα χρήματα τα οποία λείπουν ή δημιουργούν πρόβλημα δεν αναφερόμαστε τουλάχιστον ε, στα, ε, ε, στους πόρους ευρωπαϊκούς. Χρειάζονται επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, αλλά για να έχουμε καλή χρηματοδότηση χρειαζόμαστε καλό σχεδιασμό, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι μπορεί να γίνει κατά την άποψή σας για αυτό το θέμα. Τρίτον, επανειλημμένα έχουμε διαπιστώσει ότι όταν χρειαζόμαστε πληροφόρηση, ε, ζητάμε πληροφορίες και όταν λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές, ξεκινούμε από την αρχή ότι γίνονται σεβαστά ε, γίνονται σεβαστές οι διατάξεις από τις ε, χώρες μέλη και τελικά καταλήγουμε να γυρίζουμε γύρω-γύρω από το ίδιο θέμα χωρίς να μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι αναφορές ε, καταδεικνύουν σαφώς ότι και οι χώρες μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ε, όσον αφορά το θέμα αυτό. Εμείς ξεκινάμε πάντα από την αρχή ότι οι νόμοι είναι αρκετοί, αλλά τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν αρκούν καλοί νόμοι. Ο κύριος Μπολάν. Ευχαριστώ. Ε, θα προτιμούσα να απαντήσουν πρώτα οι εμπειρογνώμονες και μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, οπωσδήποτε η διαπαιδαγώγηση του κόσμου θα πρέπει ε, να γίνει και θα πρέπει να γίνεται από, ε, τα, ε, από τους αρμόδιους φορείς Ε, και έτσι ώστε να μην φτάνουν όλα τα απόβλητα ε, στην αποτέφρωση και γενικώ να υπάρχει σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Ε, επομένως, ναι, σωστή εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση, αλλά από την άλλη πλευρά τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν και κάποια συγκεκριμένα μέτρα και υπάρχουν από την άλλη πλευρά και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ε, de facto ενσωματώνονται δεν θέλω να προδικάσω την ερώτησή σας, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος, την απάντησή σας, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος μας ε, είναι να έχουμε πιο δεσμευτικό, δεσμε, δεσμευτικές ας πούμε προτάσεις ε, και όσον αφορά ε, τους αποτεφρωτές και όσον αφορά περισσότερα εργαλεία και τρόπους ελέγχου, περισσότερες δυνατότητες ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζει την ε, κοινοτική οδηγία. Το λέω αυτό ε, με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και υπό την αίρεση της απάντησης των εμπειρογνωμόνων. Ο Δόκτωρ Ράιζιγκερ θα απαντήσει πρώτα. Θέλω πολύ σύντομα να απαντήσω. Ε, στην ερώτηση του κυρίου Μπάντιγκερ όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης. Ορισμένες χώρες δεν συμπεριλαμβάνονται, όπως παρατηρήθηκε σωστά, αλλά και αυτή η γενική προσέγγιση της η ιεράρχηση των αποβλήτων αυτό είναι μία προϋπόθεση ε, λόγω της, ε, του, της οδηγίας πλαισίου. Είναι μία προϋπόθεση της μεσοδολογίας. Αλλά υπάρχει και στη νέα οδηγία πλαίσιο, η οποία καθορίζει το υποχρεωτικό ποσοστό ανακύκλωσης ε, και το διαχωρισμό των αποβλήτων σε μέταλλα, πλαστικά, απόβλητα κλπ. ανάλογα με τη σύστασή τους. Αυτές είναι οι γενικές υποχρεώσεις ε, μέσω ε, των οποίων μπορούμε να κάνουμε και σωστές αναλύσεις ανάλογα με το είδος των αποβλήτων. Τώρα, η δέσμευση και η συμμετοχή της ε, κοινή γνώμης. Η έκθεση αναφέρει στις συστάσεις της ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές, οι τοπικές υπηρεσίες, ε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία συνείδηση στους πολίτες για το όλο σύστημα της ε, διαχείρισης ε, να αυξηθεί η ενημέρωση, γνώσης, πληροφόρηση για να παγιωθεί, να εδραιωθεί μία σωστή διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων. Και αυτό περιλαμβάνεται στις συστάσεις της ε, μελέτης. Ε, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις. Ε, απαντώ στην κυρία Άουκεν από τη Δανία. Από ό,τι ξέρω, για τη Δανία, η Δανία έχει ένα υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης κατασκευαστικών υλικών, ε, οικοδομικών υλικών, ε, Πολύ λοιπόν ε, υψηλό ποσοστό ανακύκλωση οικοδομικών υλικών και μπαζών. Και άλλων υλικών καταδαφίσεων. Ή ανακυκλώνεται ή αποτεφρώνονται αυτά τα υλικά. Εξαρτάται τώρα ε, σε άλλα σημεία του κόσμου τι γίνεται. Εξαρτάται και από την τιμή των πρώτων υλών μετά το 2008 έχει σημειωθεί αύξηση των τιμών ε, πρώτων υλών, οπότε πρέπει να εγγυηθούμε ότι η ανακύκλωση, η διάθεση των ε, αποβλήτων αυτών ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ο τρόπος της διαχείρισής τους να οδηγεί στο σωστό αποτέλεσμα. Εγώ δεν διαπίστωσα στην αναφορά ότι η Κομισιόν είπε ότι τα κράτη-μέλη κάναν τα πάντα σωστά. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι βασίζονται σε αυτά που τα κράτη-μέλη τους λένε. Αν αυτά που τους λένε τα κράτη-μέλη είναι συνεπή, τότε δεν έχουν λόγους αμφισβήτησης των στοιχείων. recommendations are for how to, to, to improve this implementation. Um, with respect to, I think... Όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Μπουλόν, νομίζω, Εάν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε αντίθετα, αντίστροφα και οι πολίτες να ενισχύουν τα, τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό γίνεται, διότι στην Αυστρία, στην αρχή της δεκαετίας, δεκαετίας του 90 είχαμε μια έντονη δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών. Αυτό τώρα λίγο έχει, έχει φθήνει, έχει μειωθεί. Αλλά δεδομένου ότι εφαρμόζουμε τώρα μια, ένα διαχωρισμό των αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση των ε, υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως νομικά δεσμευτικό. και προς τον κύριο Ιτουργκάης το μόνο που μπορώ να πω είναι χρειάστηκαν περίπου 5 με 10 χρόνια στη Βιέννη να δημιουργήσουμε, να, να κατασκευάσουμε έναν αποτεφρωτή αποβλήτων με την συμμετοχή και διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων. Ε, καταρχάς όμως δώσαμε βάρος στην ε, δημιουργία στο το δυνατόν λιγότερων αποβλήτων και απορριμμάτων ε, ε, καταγράψαμε όλες τις ανησυχίες, κάναμε στη διαβούλευση, ε, μελετήσαμε το, το, κάναμε μελέτη κόστους ωφέλους και αν μας συμφέρει να κατασκευάσουμε αυτό τον αποτεφρωτή. Θέσαμε στόχο χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών από ό,τι θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια και επιπλέον δαπάνες για να πείσουμε τους πολίτες μας να πει να έχουν αντίρρηση. Ο κύριος Μπολάν. Ναι, πολύ σύντομα για να απαντήσω λίγο σε αυτά που μόλις είπε ο εμπειρογνώμονας. Νομίζω ότι όσον αφορά τη διαλογή των απορριμμάτων και τη διαπαιδαγώγηση του πληθυσμού, εγώ έχω πίσω μου την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι σημαντικό είναι διαρκώς να εξηγεί κανείς στον κόσμο τι σημαίνει η επιλογή, διαλογή ε, των ε, αποβλήτων. Επίσης, ε, να του εξηγεί πόσο κοστίζει η διαλογή των απορριμμάτων σε σχέση με την τον φόρο, ο οποίος αν δεν υπάρχει διαλογή, ο φόρος για τη μεταφορά ε, και την αποτέφρωση των απορριμμάτων είναι πάρα πολύ ψηλός. Δίνοντας λοιπόν αυτό το κόστος που θα πρέπει να πληρώνουν μέσω του δημοτικού φόρου ε, και εάν εξηγήσουμε πόσο θα μειωθεί ο φόρος αυτός, αλλά και πόσο καλό θα κάνει στο περιβάλλον ε, η διαλογή των απορριμμάτων, νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαπαιδαγωγεί στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, για την συνεργασία. Βεβαίως αυτή η έκθεση θα είναι αυτή ε, η έρευνα θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο και στα χέρια του συναδέλφου Γεωργάης αλλά και όλων των συναδέλφων. Και τώρα θα περάσω αμέσως στα επόμενα ε, δύο σημεία. το σημείο 6 γιατί κάναμε μία αλλαγή στην, στην σειρά των θεμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την σταλφο Μπαλζάνη, ε, η οποία έχει έρθει εδώ για να μας βοηθήσει με τις ε, δύο ε, αναφορές που έχουμε. Έχουμε πολλούς εγγεγραμμένους αγορητές. Να δώσω λοιπόν άμεσα τον λόγο στον πρώτο από τους ε, ενδιαφερόμενους σε σχέση με αυτές τις αναφορές και να πούμε ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 5-6 λεπτά. Ε, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρενάτ Ρέπλιγκερ από το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Βολιβέ Σαλαμπέρ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Εκπροσωπώ την Ένωση Γονέων ε, του Ευρωπαϊκού Σχολείου στις Βρυξέλλες στην Βολουέ. Ε. Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν υποβάλει μία αναφορά με πάνω από 6.000 υπογραφές στις ε, αρμόδιες αρχές και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Έχουν τα σχολεία αυτά 10.000 μαθητές και ο μεγάλος αυτός αριθμός εκφράζει τις έντονες ανησυχίες των γονέων. Τα μεγάλα σχολεία στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο δεν είναι σχολεία της ε, ε, ελιτιστικά, της αφρόκρεμας δηλαδή, σε ορισμένα μάλιστα υπολείπονται των δημοσίων σχολών των κρατών μελών όσον αφορά την δυνατότητα επιλογής ε, θεμάτων και διδασκαλίας. Υποφέρουν από ανεπαρκείς υποδεμές δεδομένου ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση θέσεων και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί ένα άνοιγμα αυτού του συστήματος. Εμείς οι γονείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μελέτες ε, σκοπιμότητος, ότι ο στόχος είναι η ε, αποδοτικότητα, όμως δεν, και επίσης έχουμε υπόψη μας και την ανάγκη περικοπών. Όμως πιστεύουμε ότι αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν ε, ισόρροπα και, και συνετά και δεν νομίζουμε ότι αυτή η πρόταση αντικατοπτρίζει αυτή την επιθυμία μας. Εμείς πιστεύουμε ότι τα σχολεία αυτά, η λειτουργία των σχολείων επιδεινώνεται και η απόδοσή τους επιδεινώνεται διότι έχουν ε, υπερβολικό αριθμό μαθητών. Παραδείγματο χάρη στο Βολουέ, το σχολείο χτίστηκε για 2.400 μαθητές ενώ του χρόνου θα έχουν πάνω από 3.200 μαθητές και αυτή ο υπερπληθυσμός, αν θέλετε, ε, των μαθητών ε, θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Γενικά, τα μεγάλα σχολεία ε, χάνουν από απόψεως αριστείων και αρίστων επιδόσεων και ο μέσος όρος τελικά των επιδόσεων είναι χαμηλότερος από τα άλλα σχολεία. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες να βρούμε αίθουσε διδασκαλίες για να μπορούν να διδαχθούν όλα τα παιδιά και γίνονται μαθήματα πρωί και απόγευμα. Τώρα, οι περικοπές ε, του προϋπολογισμού θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο τις εργασίες, τη λειτουργία και την απόδοση των σχολείων. Εμείς προσπαθούμε με τα δόντια να διατηρήσουμε έναν ε, συντονισμό και μία συνοχή στη διδασκαλία, ε, όμως ε, αυτές οι περικοπές μπορεί ίσως να είναι αναγκαίες ως ένα μέσο ανάγκης αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να εδρεωθούν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Δημιουργούνται τεράστιες δυσκολίες στο διδασκαλικό πρόγραμμα και Ορισμένα μαθήματα δεν θα μπορούν να διδαχθούν. Ε, ορισμένα μαθήματα δεν μπορούν πλέον να διδαχθούν στη μητρική γλώσσα. Παραδείγματο χάρη η χημεία. Η χημεία για παιδιά με πορτογαλική μητρική γλώσσα δεν θα μπορεί πλέον να διδαχθεί στα πορτογαλικά. Και επίσης άλλα μαθήματα τελικά διδάσκονται ε, μόνο σε δύο παιδιά. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε προσοχή στα ουσιαστικά θέματα και όχι σε μεμονωμένα συμφέροντα. Στις Βρυξέλλες ο προϋπολογισμός έχει διευρυνθεί διότι το 2012 ε, θα αρχίσει η λειτουργία ενός τέταρτου σχολείου. 50% του, του, του, του αυξημένου κόστους ε, θα διατεθούν ε, από τις συνδρομές των μαθητών και 50% από το γενικό προπολογισμό της Ένωσης. Εμείς ως γονείς θέλουμε να γίνει η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών Λειτουργία ε, λειτουργίας και να μην ε, εφαρμοστεί ένας, μια γενική περικοπή των κονδυλίων χωρίς ενδελεχή εξέταση των περιπτώσεων. Από το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Ίκλου, ο κύριος Μωράν. Καλημέρα σας. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κυδεμόνων του Ευρωπαϊκού Σχολείου ε, Βρυξέλ 1, που είναι στο Ήκλο. Εκπροσωπούμε 6.000 ανθρώπους μεταξύ μαθητών, γονέων κτλ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που ασχολείται με την αναφορά μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, μια και συζητιέται ο ε, προϋπολογισμός και οι προοπτικές 13-20. και χαίρομαι που μπορούμε να μιλήσουμε για τις ανησυχίες μας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λίγο τα ευρωπαϊκά σχολεία για όσους δεν τα γνωρίζουν. Ε, υπάρχουν λοιπόν 14 σχολεία ε, τα οποία ε, υποδέχονται παιδιά των οποίων οι γονείς δουλεύουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τέσσερα σχολεία στις Βρυξέλλες, εκ των οποίων το ένα στο Ήκλο. Στο ήκλου έχουμε 3.000 μαθητές από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Λύκειο και κατατάσσονται οι μαθητές αυτοί σύμφωνα με τη μητρική τους γλώσσα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Ευρωπαϊκού Σχολείου και αυτή την ιδιαιτερότητα θα πρέπει κανείς να την κατανοήσει σαφώς. Αυτή η ιδιαιτερότητα Τη επιτρέπει να υποδέχεται το σχολείο μαθητές οι οποίοι φτάνουν ενδεχομένως στη μέση της σχολικής χρονιάς και συνεχίζουν λοιπόν ε, στην δική τους γλώσσα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα όταν λήξει ενδεχομένως το συμβόλαιο των γονέων να επιστρέψουν στην χώρα τους και να ενταχθούν στο εκεί σχολικό σύστημα. Ε, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί τα σχολεία αυτά έτσι ώστε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να στέλνει εκεί τα παιδιά του. Ε, εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου ε, πρέπει να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό και γιατί ε, ε, αφορά ένα θέμα προϋπολογισμού, αλλά και γιατί ε, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μαζί σας, για σας, οι βοηθοί σας ε, και τα λοιπά, μπορεί να στέλνουν τα παιδιά τους στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Όσον αφορά τώρα το οικονομικό πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δεταμένο ε, το 2011 είχε κάνει μια πρόταση προϋπολογισμού 271 εκατομμύρια για το 2012 Ε, και για το 12 προτείνονται 169 ε, εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός των ευρωπαϊκών σχολείων αντιπροσωπεύει περίπου το 2% ε, του διαχειριστικού κόστους και επομένως πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι τελευταίοι δημοσιονομικοί περιορισμοί που έχουν ε, επλήξει τα ευρωπαϊκά σχολεία και σας ανέφερα τα θέματα αυτά η συνάδελφός μου προηγουμένως έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα ε, στην λειτουργία τους ε, είχαν προβλεφθεί μειώσεις των μαθητών στις τάξεις και διάφορες άλλες περικοπές. Επίσης, ε, είχε, ε, ε, επομένως σαν λύση έχει δοθεί το ενδεχόμενο αύξησης των παιδιών που φοιτούν σε κάθε τάξη από 26 δηλαδή να γίνουν 28 τα παιδιά έτσι ώστε να γίνονται πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες διδασκαλίας για τους ε, διδάσκοντες. Ε, επίσης ε, θα απολυθούν κατά κάποιο τρόπο κάποιοι καθηγητές με την έννοια ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους οι οποίες λήγουν φέτος. Στα ευρωπαϊκά σχολεία παραδοσιακά δίδεται μεγάλη προσοχή σε παιδιά με ιδιαιτερότητες ε, που χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης, είτε παιδιά με κινητική αναπηρία, είτε ε, μαθησιακές ε, δυσκολίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Επίσης, η διαχείριση του ε, ωραρίου, ε, η οποία είχε προβλεφθεί έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν όλες οι δραστηριότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Εν συμπεράσματι μπορώ να πω ότι ε, η αναφορά μας εγγράφεται στην μεγάλη κινητοποίηση της 12ης Απριλίου κινητοποίηση η οποία αφορούσε όλα τα σχολεία και πρέπει σήμερα να επαναλάβουμε ότι θα πρέπει να καταβληθούν κάθε δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε ε, να συνεχίσει η λειτουργία των σχολείων αυτών. Σας διαβεβαιώ ότι κάθε ευρώ που δίδεται στα σχολεία αυτά χρησιμοποιείται με πολύ λογικό ε, τρόπο. Επομένως έχουν γίνει ήδη πολλές περικοπές, επιπλέον ε, περικοπές ε, θα ε, δημιουργήσουν πρόβλημα διαχείρισης όλου του σχολικού συστήματος. Ε, να πω επίσης ότι το 80% του προϋπολογισμού αφορά τη μισθοδοσία των διδασκόντων και επομένως το υπολείπον ποσοστό μας αφήνει πάρα πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρξουν επιπλέον περικοπές αυτές τουλάχιστον που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, να σας καλέσω καλέσω να ε, ε, επισκεφθείτε τα ευρωπαϊκά σχολεία. Πρόκειται για σχολεία που αποτελούν πρότυπο ε, και πραγματικά θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μας είναι τόσο προσφυλή τα ευρωπαϊκά σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Interparents. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι αντιπρόεδρος της οργάνωσης Interparents. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ομπρέλα, μπορούμε να πούμε, που εκπροσωπεί όλους τους γονείς των μαθητών από όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, στα οποία αναφέρθηκαν οι προλύσαντες. Το Interparents είναι ο επίσημος συνομιλητής στα πλαίσια του συστήματος θα τόσο στο Δυτικό Συμβούλιο και συμμετέχουμε και στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δίνει τη ευκαιρία να βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω μετά όσα είπαν οι προλύσαντες όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και ότι ουσιαστικά έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα τις περικοπές που γίνονται στα σχολεία αυτά. Και οι περικοπές αυτές έχουν επηρεάσει και τις μεθόδους διδασκαλίας. Γι' αυτό το λόγο είδατε και όλες αυτές τις διαδηλώσεις των γονέων τους τελευταίους μήνες. Μου ζητήθηκε να επικεντρωθώ στα δημοσιονομικά ζητήματα, στα ζητήματα προπολογισμού και ακριβώ για αυτά θα μιλήσω. Το 2011 ξεκινήσαμε άσχημα. Ο προπολογισμό εγκρίθηκε από το Δυτικό Συμβούλιο για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στη συνέχεια μειώθηκε ο αρχικός αυτός προπολογισμός κατά 7 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Και αυτό είχε να κάνει με μία απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και ως αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά σχολεία έπρεπε να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους και να κάνουν κάποιες πολύ επίπονες περικοπές όσον αφορά τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσπαθούσαν να εφαρμόσουν. Καταβλήθηκαν πολύ σημαντικέ προσπάθειε στα σχολεία αυτά προκειμένου να μην γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν συνάδει απόλυτα με το δημοσιονομικό έτος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα σχολεία να καταφέρουν να οργανώσουν σωστά την εργασία τους βάσει των περικοπών αυτών που είχαν γίνει. Ορισμένα σχολεία λοιπόν χρειάστηκε να εφαρμόσουν το σύστημα του 12 τιμωρίου και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν ήταν καθόλου θετικό και δεν βοηθά καθόλου τη δημοσιονομική διαχείριση των σχολείων. Το πρόβλημα εντάθηκε ακόμα περισσότερο με μια απόφαση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απόφαση που ελήφθη πέρυσι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να περιοριστεί η ευρωπαϊκή συμβολή κατά το 2012, κατά 1,6 περίπου εκατομμύρια. Πέρα από την απόφαση αυτή, τα ίδια τα ευρωπαϊκά σχολεία εντόπισαν επιπλέον ανάγκες οι οποίες αντιστοιχούν σε 288 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είδαμε ότι παράλληλα η κοινοτική συμβολή ήταν 179 εκατομμύρια ευρώ. Για το 2012 λοιπόν τα σχολεία είχαν να αντιμετωπίσουν μία κατάσταση περικοπών που αντιστοιχούσαν περίπου σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο για τα σχολεία να λειτουργήσουν βάσει της κατάστασης αυτής. Το τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων ευρωπαϊκών σχολείων κατέβαλαν σημαντικότερε προσπάθειε για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα αυτά και η Γενική Γραμματεία των Ευρωπαϊκών Σχολείων μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Μόνο ότι καταβλήθηκαν πολύ σημαντικέ προσπάθειε, τα σχολεία χρειάζονται ακόμα εκα... συνολικά 168 εκατομμύρια ευρώ επομένως 4 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον όσον αφορά την κοινοτική συμβολή, την κοινοτική συνεισφορά. Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε στα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούστηκαν εκεί πέρα και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω περικοπές. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός προπολογισμός για τα ευρωπαϊκά σχολεία για το 2012 βρίσκεται λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο του 2011 κατά ένα μισό εκατομμύριο περίπου, το οποίο βέβαια δεν είναι κάποιο πολύ σημαντικό ποσό. Η αύξηση είναι μικρή. Και βλέπουμε ότι η αύξηση αυτή δεν ανταποκρίνεται και στο ποσοστό του πληθωρισμού. Δεν λαμβάνει επίσης υπόψη κάποιες εξελίξεις το Σεπτέμβριο του 2012, όπως ακούσατε, θα αρχίσει να λειτουργεί και ένα τέταρτο σχολείο στις Βρυξέλλες και θα ανοίξει και ένα νέο ευρωπαϊκό σχολείο στο Λουξεμβούργο. Από το Σεπτέμβριο του 2011 θα έχουμε επιπλέον 800 μαθητές στα ήδη φυστάμενα ευρωπαϊκά σχολεία, με ένα προπολογισμό ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί καθόλου. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα 80% περικοπές, ενώ οι ανάγκες παραμένουν οι ίδιες και μάλιστα αυξάνονται. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ε, και πάρα πολλές περικοπές, οι οποίες τελικά θα γίνουν σε τομείς που θα επηρεάσουν άμεσα τους μαθητές και ακούσατε κάποια από τα παραδείγματα από τους προλύσαντες. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα ευρωπαϊκά σχολεία βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, έχει να κάνει με το ότι δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε να συμβάλλουν τα κράτη-μέλη μέσω της παροχής μισθοδοσίας για τους διδάσκοντες. Δεν έχουν καλυφθεί όλες οι απαιτούμενες θέσεις με αποσπασμένους καθηγητές, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα ίδια τα σχολεία να προσλάβουν τοπικά διδάσκοντες και πρέπει στη συνέχεια να πληρώσουν τους καθηγητές αυτούς από το δικό τους προπολογισμό, ενώ κανονικά οι θέσει αυτέ έπρεπε να καλυφθούν από αποσπασμένου καθηγητέ από τα κράτη-μέλη που θα πληρώνονταν προφανώ από τον Εθνικό Προπολογισμό αυτών των κρατών μελών. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, πριν από 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε την έκθεση BES, στα πλαίσια τη οποία υπήρχαν κάποια πολύ σημαντικά σημεία όσον αφορά τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Το 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Honeyball, η οποία συμπεριλάμβανε κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε περαιτέρω να αναπτυχθεί το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων. Βλέπουμε τώρα ότι η μεταρρύθμιση την οποία είχε ζητήσει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο εν μέρη έχει, έχει εφαρμοστεί, χωρίς να υπάρχει μια γενική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν είναι βραχυπρόθεσμες, δεν είναι σωστά προετοιμασμένες, δεν υπάρχει απαραίτητη παρακολούθηση της εφαρμογής τους Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, δεν έχει γίνει κάποια μελέτη αντικτύπου, δεν έχει γίνει μελέτη όσον αφορά το παιδαγωγικό αντίκτυπο των περικοπών αυτών, δεν έχει γίνει κάποια αξιόλογη μελέτη κόστου ωφέλου όσον αφορά τον, τον προτινόμενο προπολογισμό για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Μολονότι, όπω σα είπα, προβλέπεται μια πολύ μικρή αύξηση στον προπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε κάποιε προτάσει στο παρελθόν, το ίδιο κάνανε και οι ενώσει των γονέων οι οποίες ε, συμφώνησαν με τις ε, προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προτάσεις αυτές είχαν να κάνουν με την ε, βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στα ευρωπαϊκά σχολεία, με την πρόθεση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία αυτά. Βλέπουμε όμως τώρα ότι το ίδιο το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Σχολείου κινδυνεύει αμεσότατα. Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια και το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχές και ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου. Θέτουμε επίσης εν κινδύνο όχι μόνο το μοντέλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, αλλά και το μέλλον άλλων σχολείων. Καταλαβαίνετε ότι το Ευρωπαϊκό Σχολείο αποτελούσε παράδειγμα προς για πολλά άλλα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σοβαρή κοινή συζήτηση όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Οι αποφάσει αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Πρέπει επίση να αναθεωρήσει τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι από τη μια θέτει κάποιε προτεραιότητε όσον αφορά το προσχέδιο προπολογισμού για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Εμείς όμως θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση θα πρέπει να παγώνει ο προπολογισμό των σχολείων αυτών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκθεση Hannibal και γενικότερα προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που γίνανε το 2005. Ολοκληρώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν πιστεύουμε ότι το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Σχολείου είναι κάτι το εντελώ θεωρητικό και το αφηρημένο. Είναι κάτι το οποίο βιώνουν τα παιδιά μα σε καθημερινή βάση. Είναι κάτι το οποίο είχαν προωθήσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον δημοσίω. Μάλλον ζητάμε από εσά, του Ευρωβουλευτέ, να προασπίσετε τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Σχολείων, να προσπίσετε το ίδιο το μοντέλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, να έχετε μια επικοδομητική προσέγγιση στον τομέα αυτό. Και θα θέλαμε επίση να σα επενθυμίσουμε ότι την Πέμπτη του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα ψηφίσει την έκθεση Καβαντά για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Η έκθεση αυτή υπεραμείνετε των προσδοκιών μας και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε λοιπόν να λάβετε υπόψη σας πολύ σοβαρά την αναφορά μας αυτή όταν θα ψηφίσετε για την έκθεση Καβαντά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μέσα στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ε, εάν δεν κατάλαβα καλά και η Ρενε έχει ζητήσει το λόγο ξανά. Ευχαριστώ. Α, ναι, είμαι η Γενική των ε, Ευρωπαϊκών Σχολείων. Δεν ζήτησα το λόγο, αλλά αφού ε, μου τον δίνετε, ευχαρίστως να μιλήσω. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τους γονείς, ε, τους εκπροσώπους των γονέων δηλαδή και αυτά που είπαν. Θα ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα και να προσθέσω και κάποια άλλα γιατί δεν συμφωνώ και με όλα όσα υπόθηκαν. Είναι γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία ε, έχουν χρηματοδότηση και από τα κράτη-μέλη ε, μέσω της απόσπασης καθηγητών είναι γεγονός ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα ε, μετά τη διεύρυνση και τον ε, υψηλό αριθμό ε, των μαθητών κυρίως στις, στους τομείς των κεντρικών γλωσσών είναι γεγονός έλεγα ότι χρειάζονται πολλές αποσπάσεις καθηγητών και πραγματικά αυτό δημιουργεί δημοσιονομική δυσκολία. το Ανώτατο Συμβούλιο ε, και μετά από τη συστάση του Κοινοβουλίου ε, έχουν ε, γίνει δεκτά κάποια πράγματα και μετά τα ψηφίσματα του 2002 και του 2005 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μεταρρύθμισης και της χρηματοδότησης και της διακυβέρνησης ε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα συμφωνήσω με τους γονείς. Ε, έχουμε κάνει προτάσεις όσον αφορά την κατανομή ε, των βαρών, έτσι ώστε να κατανεμηθούν καλύτερα τα βάρη. Βεβαίως δεν επιτύχαμε όλα αυτά τα οποία ζητούσαμε. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή 64 θέσεις ε, επί 1512 που δεν έχουν καλυφθεί από τις χώρες μέλη. Είναι γεγονός ότι έχουμε το πρόβλημα αυτό. Άλλες πηγές ε, χρηματοδότησης ε, είναι από την ε, εισφορά των γονέων στην κατηγορία 3. Όμως στην κατηγορία 3 έχουμε όλο και λιγότερα παιδιά γιατί είναι τόσο πολλές οι αιτήσει για την κατηγορία 1 και για τις Βρυξέλλες και για το Λουξεμβούργο που δεν παραμένουν θέσεις για την κατηγορία 3. Έχουμε επίσης την ε, συμβολή της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, που γίνεται βάση της σύμβασης που υπάρχει στα, στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Το 2012 θα ανοίξουμε τις Βρυξέλλες 4 και άλλο ένα σχολείο. Ε, και είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός μας είναι μάλλον περιορισμένος και πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγάλες ε, προσπάθειες ε, σωστής διαχείρισης. Επίσης, το ανώτερο συμβούλιο μας, έχουν, μας έχει ζητήσει να λάβουμε διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε να ελέγχουμε τον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών σχολείων μεταξύ των οποίων μείωση ε, των ε, αποδοχών των διδασκόντων που μπορεί να φτάσει στο 20 και στο 30% και αυτό θα μας δημιουργήσει πρόβλημα γιατί κάποιες χώρες δεν βρίσκουν πλέον καθηγητές ε, που να δέχονται να αποσπαστούν στα ευρωπαϊκά σχολεία λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των ε, ε, αποδοχών. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί πολύ τους γονείς είναι η αναθεώρηση των αποφάσεων του Ανώτερου Συμβουλίου όσον αφορά την δημιουργία τάξεων και ομάδων ε, εκπαίδευσης. Πρέπει να πω ότι σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν γίνει και μετά από σημαντικές συζητήσεις που έγιναν και στην Παιδαγωγική Επιτροπή και στη Δημοσιονομική Επιτροπή αλλά και στο Ανώτερο Συμβούλιο, κάποια μέτρα ε, αμβλήνθηκαν ε, σημαντικά. Και ε, υπάρχει πρόβλημα ακόμα για ένα μικρό αριθμό μαθητών, πέντε μαθητές συγκεκριμένα. Είναι γεγονός ότι ζητούμε ε, εξορθολογισμό από πλευράς ε, των σχολείων. Όσο γίνεται περισσότερο εξορθολογισμό, έτσι ώστε ε, τα κυριότερα στοιχεία να προσφέρονται στους μαθητές μέσω ομαδοποιήσεων διαφόρων επιπέδων ή μέσω ομαδοποιήσεων ε, μαθητών από διαφορετικούς ε, ε, γλωσσικούς τομείς έτσι ώστε να τους προσφέρετε, να τους παρέχετε η διδασκαλία στις κεντρικές γλώσσες, αυτές που εμείς ονομάζουμε Lang véhiculaire τις κεντρικές γλώσσες πράγμα που θα επιτρέψει σε μαθητές να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να γίνουν δίγλωση. Για να επανέλθουμε στα δημοσιονομικά, είναι γεγονός ότι το 2011 ε, είχαμε μία περικοπή της τάξης των 15 εκατομμυρίων και επομένως ε, με μεγάλη προσοχή θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά. Έχουμε περικόψει επίσης ε, πολλές διοικητικές δαπάνες από τη Γενική Γραμματεία. Ε, πρέπει να πω επίση ότι προσπαθήσαμε να μειώσουμε όσο γίνεται λιγότερο τις παιδαγωγικέ δαπάνες και προσπαθήσαμε να βρούμε χρήματα, να αντλήσουμε πόρους από άλλους κλάδους ε, κάποιους εξοπλισμούς ας πούμε, των σχολείων που δεν έπρεπε ε, επιγόντως να αντικατασταθούν ή να ανακαινιστούν ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην μειώσουμε τις παιδαγωγικές δαπάνες. Βεβαίως έχουμε επίγνωση des difficultés économiques dans tous les États membres. Ε, ε, έχουμε πλήρη επίγνωση της ειδική οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη. Μην ξεχνούμε ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία ε, είναι μια διακυβερνητική, ένας διακυβερνητικός οργανισμός που διέπεται από τις 27 χώρες μέλη ε, και επομένως ε, και οι χώρες μέλη ελέγχουν αυστηρά τα, τον προϋπολογισμό και την χρήση των πόρων τόσο αυστηρά όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς καταβάλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να προσφέρουμε στα παιδιά και στους μαθητές το καλύτερο επίπεδο διδασκαλίας και δεν θέλω να ακούω ότι ε, θα μειωθεί δραστικά το επίπεδο διδασκαλίας ε, ή ότι έχει ε, μειωθεί το επίπεδο διδασκαλίας. Αυτό δεν είναι αληθές. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά ας πούμε το απολυτήριο των μπακαλωρεά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά παίρνουν τον μπακαλωρεά και όλο και καλύτερους βαθμούς επιτυγχάνουν τα παιδιά αυτά. Επίσης έχουμε ένα σχολείο ε, το οποίο ελέγχεται βάσει της ε, συμφωνίας της ε, Πίζας και πραγματικά τα σχολεία μας είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, ειδικά το Λουξεμβούργο 1, είναι από τα καλύτερα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη και την Κορέα και την Κίνα, βάσει του ελέγχου των σχολείων. Γι' αυτό λοιπόν ας μην δραματοποιούμε τα πράγματα. Βεβαίως εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ειδική το, τον ειδικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών σχολείων, ε, την, δυνατότητα διδασκαλίας αποκλειστικά στη μητρική γλώσσα ή και στη μητρική γλώσσα των παιδιών. Ε, θα ήθελα να τελειώσω ε, και ε, λέγοντας το ίδιο που ε, ζήτησε και ο εκπρόσωπος των γονέων, ο κύριος Σορέν, δηλαδή να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να μην μειώσουν στον προϋπολογισμό κεφάλαιο 5, να μην μειώσουν τους πόρους για, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για, συγγνώμη, για τα ευρωπαϊκά σχολεία. ευχαριστώ πολύ. η πρόεδρος η συνάδελφος Φρανσίσκα Παλτζάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είχε, ε, ε, είχαν όλα αυτά τα οποία ακούσαμε ε, γιατί με τον τρόπο αυτό κατανοούμε το ευρωπαϊκό πνεύμα και το πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά σχολεία και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικότερα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό το οποίο αποτελεί πλέον και συγκεκριμένο κεφάλαιο του τριμερούς διαλόγου. Ε, ακριβώς δηλαδή στο νέο τριμερή διάλογο εμείς έχουμε ε, προβλέψει έναν, ε, μια ειδική παράγραφο για τον σωστό και δόκιμο, σωστή και δόκιμη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων. Αυτό βεβαίω είναι ένα όρο ο οποίος μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Αλλά εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τροποποίηση του αριθμού των μαθητών. Ε, τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τον προπολογισμό. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη διαδικασία. Έχει ξεκινήσει η ανάγνωση στις μόνιμες αντιπροσωπείες, τα κορεπέρ. Ε, γίνεται βεβαίως προσπάθεια να μειωθεί μέχρι το μεδούλι, λέει η ομιλήτρια, ο προϋπολογισμός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί να μην υπάρξουν τουλάχιστον περικοπές. Ε, ήθελα να πω ότι μετά τον Ιούλιο θα γίνει η επίσημη πρώτη ανάγνωση, ε, θα κάνει την πρότασή του το Κοινοβούλιο, θα δει τις τροπολογίες οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει έτσι ώστε ο προϋπολογισμός 2012 να σέβεται τις προτεραιότητες τις οποίες ήδη εμείς ε, υπογράψαμε τον ε, ε, μήνα Μάρτιο και ελπίζω, εύχομαι το θέμα των ευρωπαϊκών σχολείων να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο. Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ακόμα και για θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή και γενικώ πολλά ευαίσθητα θέματα. Äh, äh, Ευχαριστώ τους αναφέροντες και συμφωνήσαμε στην Επιτροπή να χειριστούμε την αναφορά αυτή ως κατεπίγουσα, διότι θεωρούμε και το αίτημα ως κατεπήγον και σημείωσα το βασικό ερώτημα. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών σχολείων. Τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ένα δημιούργημα, ένα τέκνον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα υπέρ και τα κατά του το σύστημα αυτό. Η χρηματοδότηση είναι περίπλοκη διότι είναι διτή. Δίνουν οι προπολογισμό της Ένωση, δίνουν και οι ενδιαφερόμενοι γονεί, αλλά αυτό ήταν και ο στόχο εξ αρχή. Η βασική επίκριση για μένα και εκεί συμφωνώ με τους αναφέροντες είναι η εξής. Ε, όταν μιλάμε για σχολεία, για σχολική εκπαίδευση και λέξη πολλαπλώς ότι το 80% είναι το κόστος του προσωπικού αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντοτε είναι δυνατό να γίνει μια πιο αποτελεσματική ε, χρήση του προσωπικού. Μπορούμε να που δούμε αν θέλουμε περισσότερους μαθητές, αν χρειαζόμαστε όλους τους καθηγητές, το διδασκαλικό προσωπικό δηλαδή, αν μπορούν να γίνουν περικοπές εκεί, αν μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση. Αλλά το, τα έξοδα του προσωπικού, του διδασκαλικού προσωπικού δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλά και δεν ε, υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Χρειαζόμαστε χρόνο. Το ερώτημα όμως είναι, θέλουμε τα σχολεία αυτά. Κανένας δεν έχει πει μέχρι τώρα ότι δεν θέλουμε να έχουμε τα ευρωπαϊκά σχολεία. Βεβαίως, όταν μιλάμε για μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική δομή, όλα αυτά μπορούν να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων. Όμως, ε, τα, σχολεία αυτά, τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσει και ιδιαίτερες υποχρεώσεις, ε, πρέπει να απ' τη μία να αυξήσουν τα δίδακτα, δεδομένου ότι έχουν αυξημένες δαπάνες, και αφετέρου να συμμορφωθούν με τις περικοπές. Συμφωνώ λοιπόν με τους αναφέροντες. Πρέπει να προσέξουμε ότι τα σχολεία λειτουργούν διαφορετικά από ότι οι προπολογισμοί. Οι προπολογισμοί λειτουργούν βάσει του οικονομικού έτου και τα σχολεία βάσει του σχολικού έτου. Άρα λοιπόν, οι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού του δικού μας λαμβάνονται στο μέσον της σχολικής περίοδου, της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, 80% δαπάνες ε, διδασκαλικού προσωπικού, 20% διοικητικές δαπάνες. Τώρα, μπορούμε βεβαίω να αναβάλουμε επενδύσεις ε, οι οποίες είναι απαραίτητες, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν αργά ή γρήγορα. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπολείπονται τα ευρωπαϊκά σχολεία της προόδου που γίνεται γενικώ στο εξωτερικό περιβάλλον. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε πρέπει να κάνουμε και τις απαραίτητες προσαρμογές στι υποδομέ. Λοιπόν, όταν κάποιο λέει, ε, αυτή τη στιγμή ίσω είναι η Κομισιόν, ε, ότι πρέπει να οργανωθούν τα σχολεία αυτά πιο αποτελεσματικά, πρέπει να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να δεχθούμε ότι τα σχολεία έχουν, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τα, τις πάγιες δαπάνες. Έχουν πάγιες δαπάνες τα σχολεία. Γι' αυτό ε, ζητώ να διαμορφώσουμε μία στρατηγική κατάλληλη ε, και να μελετήσουμε λεπτομερώς όλες τις πτυχές λειτουργίας των σχολείων ώστε να διαπιστώσουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι κοιτάξτε με, αυτό το, με αυτά που ζητάμε ε, θα λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία. Δια, ε, σημείωσε επίσης ότι όλα τα σχολεία δεν είναι στο Λουξεμβούργο, Στρασβούργο και Βρυξέλλες μόνο. Όλα μπορούν να συζητηθούν, Όλες τις προτάσεις μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ένα δημιούργημά μας, ε, δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τον ε, τομέα αυτόν. Ε, το δημιούργημά μας αυτό. Είναι παιδί μας τα ευρωπαϊκά σχολεία. Θα φροντίσουμε λοιπόν καταρχάς να μελετήσουμε τι περικοπές προτείνονται Εν συνεχεία θα ζητήσουμε την εκπόνηση μιας λεπτομερούς μελέτης η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλο το δημιούργημα αυτό και τους στόχους και την πορεία των ευρωπαϊκών σχολείων και τρίτον θα βρούμε τα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Τη χρηματοδότηση του θεσμού αυτού δεν είναι δυνατόν να αναγραφεί στο προπολογισμό ένα κονδύλι για τα ευρωπαϊκά σχολεία, μετά να το διαγράψουμε με ένα μολύβι και να ε, συνεχίσει να λειτουργεί ο θεσμός ε, σωστά. Αυτά δεν γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βελτζάνη, η οποία πρέπει να φύγει και θα δώσω το λόγο στον Σεραφή Τουργκάης. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι γενικά συμφωνούμε. Και η κυρία Μπαλτσάνη η οποία έφυγε δυστυχώς, δεν μπορεί να παραμείνει. Όλοι συμφωνούμε ότι τα σχολεία πρέπει να διατηρηθούν εν ζωή, βεβαίως. Όμως, δεν πρόκειται εδώ μόνο για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων. Βεβαίως χρειάζονται τις πιστώσεις και τη χρηματοδότηση. Όμως χρειάζονται επίσης και μια εξασφάλιση ποιότητας, ε, παιδαγωγικής ποιότητας. Ε, δηλαδή χρειάζονται το σωστό διδασκαλικό προσωπικό, το σωστό παιδαγωγικό προσωπικό, ε, τη δυνατότητα ε, εκπαίδευσης παιδιών με ε, ειδικέ ανάγκες, τη δυνατότητα διδασκαλίας παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες, την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεως, εδώ πρόκειται για την ε, μόρφωση νέων ε, ατόμων, νέων ε, παιδιών. Και πέραν αυτό που είπε ο κύριος Γιά, νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να συντάξουμε μία επιστολή προς τον αρμόδιο επίτροπο και να του εξέσουμε τις θέσεις μας ως Επιτροπή Αναφορών και ως θέση του Κοινοβουλίου, ώστε ο Επίτροπος ε, να γνωρίζει ε, ότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε μια επαρκή χρηματοδότηση, όπως είπε η κυρία Μπαλτσάνη, ε, για την σωστή λειτουργία των σχολείων αυτών και την εξασφάλιση της αναγκαίας παιδείας των παιδιών αυτών, της αναγκαίας μόρφωσης. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη, ιδιαίτερα στο σημείο που ζήτησε την, ε, ε, ε, μία μελέτη, σύνταξη μιας ενδελεχούς μελέτης ε, εγώ ήμουν ε, καθηγήτρια στο παρελθόν. Δέχομαι ότι θα πρέπει να γίνουν ε, ορισμένες περικοπές, αλλά παιδαγωγικές περικοπές είναι αδιανόητο. Πώς είναι δυνατόν να περικόψουμε τη μόρφωση, πώς είναι δυνατόν να περικόψουμε πτυχές της παιδείας που θα λειτουργήσουν αρνητικά στα παιδιά και ιδιαίτερα εν ώψη της Ευρώπης του 2020. Δηλαδή θα, θα δημιουργήσουμε θα εφαρμόσουμε θεσμικές περικοπές οι οποίες θα λειτουργήσουν εναντίον των παιδιών μας. Βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Γιάρ, χρειαζόμαστε μία σωστή μελέτη για να δούμε πού μπορεί να γίνουν σωστές οικονομίες, αλλά όχι πάνω στις πλάτες των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάλκομ Ρίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Οι δύο αναφορές που συζητώνται σήμερα εμπίπτουν στην προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ως σύγχρηματοδότου. Πρώτον, Εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπήρξαν και για σειρά ετών δεν υπήρξε μείωση του προϋπολογισμού λειτουργίας των ευρωπαϊκών σχολείων. Όμως, είναι γεγονός ότι κυρίως για το προϋπολογισμό του 2011 η αύξηση της τάξης του 11,5 η οποία προεβλέπεται δεν επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον στο βαθμό που ε, επιθυμούσαν τα σχολεία. Υπενθυμίζω ότι τον Απρίλιο του 2010 το Ανώτερο Συμβούλιο ε, των Σχολείων με θετική ψήφο της Επιτροπής είχε, είχαν ε, υπογράψει τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό της τάξης των 171 εκατομμυρίων όμως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Σουηδία, τέσσερις χώρες ε, και η ε, Επιτροπή ε, στο τελευταίο, στην τελευταία συζήτηση του προπολογισμού είπαν ότι ναι, μεν εγκρίνεται ο προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσει, κυρίω όσον αφορά τρία στοιχεία. Το διδακτικό προσωπικό, η διαχείριση των ε, των μαθημάτων και ένα τρίτο. Πρώτον, ο τρόπος μισθοδοσίας και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού βασίζεται ε, στον τρόπο μισθοδοσίας των ε, υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2004 υπήρξαν τροποποιήσεις κυρίως όσον αφορά τους ε, νέο εισαγόμενους ε, στο σύστημα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επομένως από τη στιγμή που υπάρχει παραλληλισμός ανάμεσα στα δύο καθεστώτα οπωσδήποτε θα έπρεπε να διευθετηθεί η διαφορά που προέκυπτε και επομένως θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί το σύστημα μισθοδοσίας ε, των ε, διδασκόντων στα ευρωπαϊκά σχολεία ε, προς το σύστημα μισθοδοσίας των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά αναλογία δηλαδή να υπάρξουν περικοπές με μειώσεις της τάξης του 15 μέχρι 21% κυρίως για τους νέους εισερχόμενου. y a un parallélisme entre les deux euh, figures professionnelles, entre les professeurs des και επίσης θα, υπήρξε και, θα υπήρχε και η απαραίτητη προσαρμογή των αποσπασμένων και των μονίμων ε, καθηγητών. Επίσης, όσον αφορά την ε, ε, δημιουργία ε, κατεπιλογής μαθημάτων είναι γεγονός ότι αυξήθηκε ο ρυθμός των απαιτουμένων μαθητών έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ειδικό κατεπιλογή μάθημα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές κάθε χρόνο οδηγούν σε μία μείωση του πραγματικού κόστους των σχολείων. Ε, και προκύπτει ένα σύστημα βάσει του οποίου η αγοραστική δύναμη των σχολείων είναι ψηλή. Αναφέρομαι εδώ ε, για, ε, αναφέρομαι εδώ σε 4 εκατομμύρια ε, σωρευθέντων κεφαλαίων που προκύπτουν και από την μισθολογική διαφοροποίηση και από την αποταμίευση. Και επομένως για το 11-12 η πραγματική περικοπή είναι περίπου στο 1, Αυτά για να ξαναθυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει όσον αφορά τα μέτρα τα οποία και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ζήτησαν ε, να λάβει ε, το Ανώτερο Συμβούλιο και το οποίο Ανώτερο Συμβούλιο έκανε δεκτές τις προτάσεις αυτές. Le budget de 2011, donc de l'année en cours. Προϋπολογισμός 2011, δηλαδή τρέχοντος έτους. Ε, αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω μείωσης. Και επομένως από τα 171 εκατομμύρια έφτασε η Κομισιόν ε, στο ποσό των 164 εκατομμυρίων. Ε, ε υπενθυμίζω ότι η αύξηση είναι της τάξης του 6,5% ενώ ο αριθμός αύξησης των μαθητών είναι 3,5% και του προπολογισμού της Επιτροπής η αύξηση είναι 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αύξηση για τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι πάρα πολύ ψηλή και ξεπερνάει κατά πολύ τον αριθμό των ε, μαθητών που φοιτούν στα ευρωπαϊκά σχολεία όσον αφορά τώρα το έτος 2012. Είναι γεγονός ότι τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια ε, ζήτησαν 169 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, το, το αίτημά τους δεν έγινε σε καμία στιγμή δεκτό στο σύνολό του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πάρει ακόμα τελικές αποφάσεις, ε, βέβαια, όμως έχει καταδείξει βάσει και της ε, θέσεως που έχει λάβει συστηματικά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον προπολογισμό 2012, δηλαδή ότι θα πρέπει να μην υπάρξουν αυξήσεις ε, σε αυτό το προϋπολογισμό. και επομένως η Κομισιόν θεωρεί ότι τα 164 εκατομμύρια δεν θα πρέπει να αυξηθούν. υπευλήθη από τη Γενική Γραμματεία των Σχολείων ε, ένας προπολογισμό της τάξης των 165,4 εκατομμυρίων, δηλαδή αύξηση λιγότερο από 1% και επομένως η Κομισιόν έκανε δεκτή την αίτηση αυτή ε, και ε, προσδοκούμε θετική ψήφο και της αρχής του προϋπολογισμού. Θα υπάρξει πάντως, όπως αναφέρθηκε, μάλλον έχει υπάρξει και μία ε, μελέτη ε, σχετικά με τον εξορθολογισμό των ε, πόρων και την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων. Έγινε προσπάθειες λοιπόν εξοικονόμησης προς κάθε κατεύθυνση με κύριο μέλημα την διατήρηση του σχολικού προγράμματος που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει απαράλλαχτο. Les, euh, et donc, nous demandons à le... Και εν πάση περιπτώσει ζητούμε από την αρχή του προϋπολογισμού να εγκρίνει αυτόν τον τελικό προϋπολογισμό που προτείνεται 165,4 εκατομμύρια για το 2012. Όσον αφορά την ποιότητα, γιατί και η Γενική Γραμματέα των Σχολείων ε, αναφέρθηκε στην ποιότητα διδασκαλίας. Αυτή η ποιότητα διδασκαλίας στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ υψηλή και η Γενική Γραμματέας αλλά και ε, ο εκπρόσωπος ε, των διευθυντών των σχολείων μας διαβεβαίωσε στην τελευταία συνάντηση ότι δεν υπάρχει κανένας ε, κίνδυνος μείωσης της ποιότητας της διδασκαλίας και του επίπεδου διδασκαλίας των σχολείων. Αυτά είχα να σας πω, με λίγα λόγια. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που συνοπτικά ήθελα να κάνω ε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θέλουν μήπως οι αναφέροντες να κάνουν κάποια τελικά σχόλια. Όχι από ό,τι φαίνεται. Όχι. συνάδελφε, θέλετε το λόγο. Ε, εντάξει, ο συνάδελφος Γιάννα παρακαλώ. Da äh, Ναι, πιστεύω και εμένα στην απόψή μου ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής Δύο, δύο συστήματα εφαρμόζονται, δύο τρόποι υπάρχουν να γίνουν περικοπές στα σχολεία και εγώ δεν δέχομαι το τόνο ούτε Ή θα περικόψουμε τους μισθούς του προσωπικού ή θα αυξήσουμε τα δίδακτα. Ε, δεν είναι μόνο λοιπόν το οικονομικό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και την υπερφόρτωση των σχολείων αυτών ε, με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, επίσης τις πολυπληθείς τάξεις που δημιουργούνται Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο πρέπει να ξέρουμε προς τα πού πορευόμεσα, πού θέλουμε να καταλήξουμε στο ταξίδι αυτό, να μελετήσουμε με προσοχή τις ανάγκες που, με, τη μελέτη αυτή που προτείνω και επίσης το προσωπικό το οποίο αυτή τη στιγμή προσλαμβάνεται σε χαμηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας ε, ναι μεν προσλαμβάνονται σε χαμηλότερη θέση, αλλά όσοι είναι πιο ψηλά από πάνω θα προχωρήσουν στις προαγωγές τους. Και αυτό πρέπει να μελετήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε με πολύ προσοχή τους λογαριασμούς και να εξασφαλίσουμε μία σωστή, ενιαία και συντονισμένη στρατηγική μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών σχολείων. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Γιάρ. Επομένως, προτείνουμε να, να προχωρήσουμε ε, την συνεργασία κυρίως με τον Επίτροπο Σεφκόβιτς στον οποίο θα αποστείλουμε ένα υπόμνημα ως Επιτροπή έτσι ώστε να του εκθέσουμε στην θέση όλα όσα διαδραματίστηκαν εδώ σήμερα και κυρίως για να επιμείνουμε να μην έχουν οι περικοπές οποιαδήποτε επίδραση ή επίπτωση στο επίπεδο διδασκαλίας. Όπως είπε και η κυρία Μπαλτζάνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έρθουμε και σε επαφή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω τους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής σε σχέση με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει σε λίγο στους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε ε, να δώσουμε στην παράγραφο που αναφέρεται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Μπαλτσάνη, να ε, δώσουμε, λέω, στην παράγραφο αυτή μία διαφορετική χρηματοδοτική κατεύθυνση. Αν δεν ε, ζητά κάποιος άλλος το λόγο, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες που ήταν παρόντες. Ευχαριστούμε τους ε, βουλευτές. Θα ε, σταματήσουμε, θα διακόψω για λίγο μάλλον τις εργασίες της Επιτροπής μας, γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι την αίθουσα. Έχουμε συνάντηση των συντονιστών.